ψηφίζουμε τροπολογία 5 με ονομαστική ψηφίζουμε. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Διανατάσσεως ισχυρός πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ονομαστική. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας.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 Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 με ονομαστική ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας ε, C, γραμμά C υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας D, αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3, Μενομαστική. ονομαστική. Έναρξης ψυχορίας Πέρας. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας J, αρχικό κείμενο, δυνατάσεως υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται εκτιμώντας και αρχικό κείμενο διανατάσεως υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το ψήφισμα το συνόλο του με ονομαστική ψηφίζουμε πέρας ψηφορίας εγκρίνεται διαδικαστική παρέμβαση Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η είπε Κοινοβουλή δεν είναι αποδεκτές ε, οι δηλώσεις όσον αφορά τα κατεπήγοντα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον κανονισμό για αυτό. Είναι κάτι απαραίτητο να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Γιατί έχουμε ένα ονομαστικέ πληροφορίε. Και έτσι οι βουλευτέ δεν μπορούν να πούνε τι σκέφτονται, τι πιστεύουν με την ε, δήλωση, την επεξήγηση ψήφου μετά το υπέρ και το κατά. Αλλά νομίζω επομένω ότι θα πρέπει όλοι μα να ξεσηκωθούμε, να διαμαρτυρηθούμε για αυτή την αδικία. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Θα πρέπει να επιτρέπονται οι επεξηγήσει ψήφου. Όπω ε, μόλι είπατε, Πρόκειται για άρθρο του κανονισμού. Σημειώνουμε πάντως την αντίρρησή σα και παίρνουμε στο ψήφισμα για τη Μαυριτανία. Ένα ψήφισμα επί του συνόλου. Διανατάσεως υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και παίρνουμε στο ψήφισμα για το Σουδάν. Κοινό ψήφισμα 7 πολιτικών ομάδων. Ξεκινούμε τροπολογία 1, ανάταση υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα επί του συνόλου με γη. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και περνούμε στην πρόταση ψηφίσματος από 92 βουλευτές mm. επί του μηχανισμού mm. γενικευμένων δεσμολογικών προτιμήσεων. Τροπολογία 1. Με ανάταση υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επί του συνόλου θέλουμε ειδική πλειοψηφία, ονομαστική ψηφορία, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Εγ... Με συγχωρείτε. Όχι. Ε, δεν εγκρίνεται. Θέλουμε ειδική πλειοψηφία. Δεν εγκρίνεται λοιπόν. Επόμενο. Πρόταση ψηφίσματος για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό, το εξηγένσης, ονομαστική, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Επιτρέψτε μου